Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι. Τα πρακτικά τη χτεσινή συνεδρίαση και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι στη διάθεσή σα. Υπάρχουν αντιρρήσει.